So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf hier Ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα την συνεδρίασή μας και πρώτα ρωτώ αν έχετε προσθήκες ή σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Άρα γίνεται δεκτή, εγκρίνεται δηλαδή η ημερήσια διάταξη. Έχω τώρα ορισμένε ανακοινώσει να μου επιτρέπετε. Θα σας τα πω μάλιστα στα αγγλικά και βέβαια θα εγγραφούν και στα πρακτικά. Πρώτα έχουμε τριμερή διάλογο για τα δικαιώματα των μετόχων με επικεφαλή στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αλλά και κάποιες αρμοδιότητες της Επιτροπής Οικονομικών σύμφωνα με το ε, άρθρο του κανονισμού υπαριθμών 54. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 27 Δεκάτου παρουσία του George Friedel της ε, Λουξεμβουργικής Προεδρίας και της Αρμοδίας Επιτρόπου και από το Κοινοβούλιο κ. Λούντζιξον με στόχο να τοποθετηθούν τα θεσμικά όργανα για βασικές πτυχές της προτάσεως και να εντοπίσουν θέματα όπου πρέπει να διεξαχθεί προόδος πριν από τον επόμενο πολιτικό τριμερή διάλογο. Θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ταυτοποίηση των μετόχων, διαφάνεια, διαφάνεια των διαχειριστών ε, περιουσιακών στοιχείων και εκεί πάλι συντρέχουσα αρμοδιότητα σύμφωνα με το 54 εκθέσεις αναχώρα και διαφάνεια των αποφάσεων tax ruling. Θα συνεχιστεί η εργασία στο τεχνικό επίπεδο και ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο τριμερή διάλογο. Επόμενο τριμήρι διάλογο για τον κανονισμό benchmark, όπου έκτος έγινε στις 28 Δεκάτου 2015 στη βάση προτάσεως για κανονισμό benchmark. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η ταξινόμηση των benchmark ως κρίσιμα σημαντικά και λιγότερο σημαντικά και το καθεστώς που θα αποδίδεται σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αυτές, ρυθμιζόμενα δεδομένα, benchmark και οι ε, σχετικές ρυθμιστικές αρχές. Το Κοινοβούλιο κατέθεσε τα βασικά στοιχεία μιας ενδεχόμενης συμβαστικής προτάσεως και ζήτησε από την Προεδρία του Συμβουλίου να επανέλθει. Επόμενος τριμηρής διάλογος προβλέπεται για τις 24 ενδεκάτου φέτος. Και έχω τώρα ανακοίνωση για μια σύνοψη αποφάσεων και συστάσεων στην συνάντηση των συντονιστών της 28 Οκτωβρίου όπου αποφασίστηκε ότι το επόμενο θέμα θα συζητήσει θα συζητηθεί μάλλον για την ε, ε, Σύμβαση φερογκαιότητας 2, Solvency 2. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας διαβάσω όλα αυτά τα νούμερα. Γνωρίζετε τι ε, θα πει Solvency 2. Οι συντονιστές της ΕΚΟΝ αποφάσισαν να αναβάλουν την απόφαση για ορισμένες προτάσεις της Προεδρίας για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την απλοποίηση κλπ. Για τις απαιτήσει σόφρονος ε, διαχειρίσεως των ε, τραπεζικών και πιστοτικών ιδρυμάτων και να μην συνταχθεί γνωμοδότηση για τον ε, μηχανισμό relocation. Και ο συντονιστής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η ίδια δεν συμφωνούσε με την απόφαση αυτή. Οι συντονιστές της ΕΚΟΝ αποφάσισαν να υποβάλουν γραπτή ερώτηση για την συμπλήρωση της Οικονομικής και Ένωσης και αυτό προβλέπεται να συζητηθεί στις 17 Νοεμβρίου. Άλλες λεπτομέρειες θα σας γνωρίσει η Γραμματεία εντός των επομένων 24 ώρων. Από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ζητείται η άδεια ανάληψης ε, ε, έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας και ως αποδεκτή λύση για την αίτηση ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών προβλέπεται το άρθρο 55. Οι άλλες επιτροπές που έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν, ρωτάω πρόεδρος. Γνωρίζω βέβαια το ιστορικό γιατί ήμουν παρόν στην σχετική διάσκεψη των Προέδρων ε, των, ε, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Μπορώ να σας διαβάσω διάφορα νούμερα τώρα. 2015 B80782 from 2015 B80784 from 2015 B80824 from this year B80825 from this year B80830 from this year B80831 from this year B80869 B80871 B80882 all from this year Όλα αυτά τα νούμερα είναι του φετινού χρόνου, δηλαδή 2015. 9 b 80900 B80908 B80911 911 good number B80912 B80916 B80919 B80938 B80974 B80981 Oh and that's it. Αυτά λοιπόν τα νούμερα και τις λεπτομέρειες θα τις δείτε στα πρακτικά εφόσον θέλετε να ανατρέξετε σε αυτά. Τώρα, για το μέλλον, εάν δεν υπάρξει ένσταση από κάποιον συντονιστή, θα συντάξει μια στάνταρδα απάντηση η γραμματεία λέγοντας ότι δεν προτίθεται ή μάλλον πρότειναν οι ε, συντονιστές να μην δοθεί συνέχεια στις αιτήσει για την ε, σύνταξη ψηφισμάτων. Αυτά λοιπόν, ακούσατε και τα σχετικά νούμερα και τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα, σημειώνει τρία της ημερησίας διατάξεώς μας που αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λίχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003-48 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ευρωπαϊκή Κοινότητα του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπομορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσει. Ο εισήγητη θα λάβει τώρα τον λόγο για να μπορέσει να εξηγήσει το κείμενό του και βεβαίως οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να σχολιάσουν. Θέλω μόνο να τονίσω ότι οι συντονιστές έχουν αποφασίσει να κατανέμονται τα θέματα αυτά, τα φορολογικά, σε μια ε, διαδοχική σειρά. Γιατί έχουμε και άλλα. Ανδόρα, Μονακό, Άγιο Μαρίνο και άλλα ε, τέτοια κράτη ε, ώστε λοιπόν κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ψάξει να βρει ποια είναι η αγαπημένη της μικρή χώρα για να κάνει τη σχετική έκθεση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταμπάτη, ο οποίος εκπροσωπεί τον εισηγητή κύριο Λούνς. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ο συνάδελφος Λούνες στέλνει, ζητά συγγνώμη που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ λόγω ήδη ανελημμένων υποχρεώσεων και προβλήματος δηλαδή στο χρονοδιάγραμμά του. Ε, ο κύριος λούνε στηρίζει τις προσπάθειες για την ε, ε, μείωση της φοροπάτης και της φοροδιαφυγής και επικροτεί τη συμφωνία με το Λιχτεστάιν για εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Ε, ως εκ τούτου, ο εισηγητής καλωσορίζει και στηρίζει την ενημέρωση και επίσης ε, προτείνει να περάσει ε, ε, σε το χρόνο ώστε να αρχίσει να ισχύει από την 1η Πρώτου 2016. Σας ευχαριστώ. Έχετε λίγο παραπάνω χρόνο αν χρειάζεστε. Όχι. Αυτά είναι, αυτά, δεν έχω άλλο κείμενο φορολόγηση των εισοδημάτων από είναι μεγάλη υπόθεση. Η παιδική μου περιφέρεια είναι γειτονική με το Λιχτεστάνι. Μπορώ να σας πω διάφορες ιστορίες για αυτή την υπόθεση. Σκιώδης ε, του ε, ΕΛΚΑ, ο κύριος Μπάλτ. Ο κύριος Μπάλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή, έστω και αν είναι απόν σήμερα, τον κύριο Σάντερ Λούνς, βρίσκω ότι είναι πολύ θετική η έκθεση του. Πρώτα η Ελβετία και τώρα το Λίχτενστάιν συμμετέχουν πλέον στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνήψε σχετική συμφωνία με το Λίχτενστάιν και είναι πολύ καλοδεχούμενη η συμφωνία αυτή διότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα κατά της φοροδιαφυγής και των απατών γύρω από τους φόρους. Η ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών ασφαλώς θα διευκολύνει το έργο των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό των φοροδιαφευγόντων αλλά και για την αποτροπή τους. Αποτροπή δηλαδή της προσπάθειας αποκρύψεως εισοδημάτων στην αλλοδαπή. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία ώστε το Λίχτενστάιν να θεσπίσει όμοιους κανόνες όπως οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι από την θέση ισχύ τη συμφωνίας του 2005 έχουν ε, επισημειωθεί σημαντικές εξέλιξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς. Για παράδειγμα η οδηγία για την δικαστική αρρωγή, για την δικαστική συνδρομή δηλαδή, καθώς και τα πρότυπα του ΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων του 2014. Ελαμβάνει μια νέα ποιότητα λοιπόν ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής με ε, το βήμα αυτό και γι' αυτό ο σκιώδης εισηγητής της ομάδας μας κύριος Ανδρέα Σβάπ συμφωνεί με τον εισηγητή κύριο Σάντερ Λούνς ότι δηλαδή θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει την συμφωνία να, μας, να με συμπαθάτε αλλά πήρα τον διπλάσιο χρόνο από τον ε, προορίσαντα κύριο Σταμπάτη και ας προσπαθήσουν οι επόμενοι να με ξεπεράσουν αν μπορούν. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ελπίζω να μην αποδειχθεί ε, η γεγονός αυτό που λέτε. Τώρα, για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μιλάμε για αυτό το όμορφο Λίχνενστάιν. Πολύ καλό σκι, ε. Λοιπόν, εκ μέρου των σοσιαλιστών και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή μας παρακολουθεί το θέμα αυτό της μείωσης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και είναι μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Φυσικά και είμαι υπέρ της απλοποιημένης διαδικασίας. Ω εισηγητή για τη συμφωνία με την Ελβετία, χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα περνάμε στι επόμενε χώρε. Τώρα το Λίχνεστάιν. Αυτό όμω που έχει περισσότερο σημασία είναι η ίδια η ουσία τη συμφωνία. Και η ουσία είναι ότι Τώρα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε καρποφόρα συνεργασία με το Λίχνεστάιν για την καταπολέμηση της φοροποφυγής και της φοροδιαφυγής. Και πρέπει να προχωρήσουμε και ακόμα πιο πέρα. Ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτόν. Θέλουμε μια συνολική συμφωνία. Θέλουμε πιο αυτόματη, αυτόματες συνθήκες για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλε χώρε και θέλουμε και περισσότερη διαφάνεια. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιλαμβάνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για κάθε νέα εξέλιξη και θεωρούμε και η σημερινή υπόθεση αλλά και άλλε παρόμοιε που θα έρθουν στο μέλλον ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Πρέπει να δράσουμε κάθε φορά που υπάρχουν παράνομε και αθέμητε φορολογικέ μεταχειρήσει. Τίποτα άλλο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που δεν παίρνετε και όλο το χρόνο που σας αναλογεί. Εκ μέρους των φιλελεύθερων δεν βλέπω εδώ σκιώδη, αλλά βλέπω την συντονίστρια. Ναι, αλλά δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω, λέει η κυρία Γκουλάρ. Ναι, αλλά για το Λίχνεστάιν εγώ ευχαρίστω να το ξαναεπισκεφθώ, λέει η κυρία Γκουλάρ, αλλά δεν θέλω να πληρώνω φόρου είναι αλλού εκτός από τη Γαλλία. Καλώ, λέει ο πρόεδρος. Σωστά. Ο Μιγγελ Ιέγκας τώρα, μέρος των Πρασίνων. Μάλιστα. Εμείς σκοπεύουμε, ε, ε, θεωρούμε μάλλον ότι είναι θετικό αυτό το βήμα, είναι ακόμα ένα βήμα το οποίο επικυρώνει τη δική μας εκτίμηση ότι δηλαδή αυτά τα σκάνδαλα που έφεραν στο δημόσιο βήμα όλη αυτή την υπόθεση ε, οδήγησαν σε μια εργασία που, στο Κοινοβούλιο που τώρα αποφέρει πια καρπούς. Ε, το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης, αυτών των σκανδάλων, του γεγονότος ότι ο, ο πολίτης δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτές οι διαφυγές ενώ οι κυβερνήσεις επιβάλλουν διαρκώς μέτρα λιτότητας, ε, βλέπουμε ότι τελικά οδήγησε σε θετικά βήματα. Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι να παρακολουθήσουμε την διαδικασία αυτή και να την αξιολογούμε. Σύμφωνα με τα όσα μπόρεσα να διαβάσω και να μελετήσω, επί της ουσίας η ανταλλαγή των πληροφοριών θα ξεκινήσει το 2016. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχουν διοικητικά θέματα, αλλά θέλουμε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση, ε, γιατί αυτό θα ήταν αρνητικό. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι Το πρόβλημα δεν λύθηκε όχι λόγω έλλειψη νομοθεσίας. Οι πληροφορίε έπρεπε να ανταλλάσσονται εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η υπόθεση με το Λιχτενστάιν επίση δεν είναι τωρινή, δεν είναι σημερινή. Υπήρξαν άλλα σκάνδαλα στο παρελθόν που όμως δεν είχαν τον αντίκτυπο που είχε το Leaks» αλλά ήδη από το 2008 υπήρχαν σκάνδαλα ανάμεσα στο Λιχτεστάιν και στην Γερμανία. Φτάσανε στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, νομοθέτησαν ε, τα θεσμικά όργανα, αλλά δεν αρκεί να νομοθετεί κανεί. Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά δεν παράγονται τα αποτελέσματα που επιθυμούμε μόνο και μόνο με την νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, να δίνεται συνέχεια και αυτόματη η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι γίνεται. Αυτό που θέλω να πω καταλήγοντας είναι ότι εδώ εμείς θα εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία που είναι θετική, αλλά ακόμη πιο θεμελιώδης είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων αυτής της νομοθεσίας, ώστε οι πολίτες να καταλάβουν πως όντως εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε, να εγκρίνουμε τη συμφωνία και πάνω απ' όλα επαναλαμβάνω, να παρακολουθήσουμε, να αξιολογήσουμε, να ζητήσουμε, να λογοδοτήσουν όλοι όσοι πρέπει να εφαρμόσουν όλα αυτά, να δούμε αν όντω εφαρμόζονται και αν μεταφράζονται σε κάτι το θετικό και το απτό για τους πολίτες. Δηλαδή, αν όντως επιτέλους ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτήσουμε την απάτη και τη φοροδιαφυγή. Σας ευχαριστώ. Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους. Σήμερα είμαστε στην 9η Νοεμβρίου. Για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το όλον αυτό 1η Ιανουαρίου 2016 θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα. Το Συμβούλιο μας έχει παρακαλέσει να εγκρίνουμε την γνωμοδότησή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή στην Ολομέλεια, την ε, μήνυ λεγόμενη Ολομέλεια τη Δευτέρα Δεκεμβρίου, ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν το ταχύτερο ε, δυνατόν. Βεβαίω, είναι προ το κοινό συμφέρον όλων των θεσμικών οργάνων η συμφωνία να προχωρήσει όσο γίνεται γρηγορότερα και να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη από τον Ιανουάριο. Και όπω εξήγησα, βρισκόμαστε ήδη στον Νοέμβριο. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό, εκτός εάν ο εκπρόσωπος του εισηγητού επιθυμεί να λάβει πάλι το λόγο. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπω κανένα να σηκώνει το χέρι. Ας κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα τεσσάρων λεπτών μέχρι ότου προσέλθει η Επίτροπος κυρία Βεστάγκερ. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να καλωσορίσω την Επίτροπο κυρία Βεστάγκερ. Έρχεται εδώ ενώπιόν μας για μια τρίτη πλέον ανταλλαγή απόψεων με την Οικονομική Επιτροπή στα πλαίσια του διασωμένου διαλόγου μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων. Από την τελευταία σας εμφάνιση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών τον Ιούλιο έχει κάνει σημαντική πρόοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του επιθετικού ε, φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων και υπάρχουν και υποθέσεις Fiat και Starbucks Αναμένουμε να μας εξηγήσετε πού βρίσκονται τα πράγματα με αυτές τις υποθέσεις και άλλα και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις και νομίζω ότι έχετε και ε, μήνυμα του ε, συναδέλφου σας Μοσκοβισή, τον οποίο είδαμε πριν από λίγο καιρό ε, για την έκθεσή μας για τις αποφάσεις τύπου tax ruling. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώσατε τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το πώς να δοθούν περισσότερες εξουσίες στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να επιβάλλουν την νομοθεσία. Η ομάδα υπηρεγνωμόνων έχει συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Λουξεμβουργικής Αρχής, Λουξεμβουργικής Προεδρίας στο ε, Στρασβούργο. Είδαμε πώς ε, συνεργάζεται η αρχή αυτή με άλλες και πώς ε, είναι οργανωμένη σε μια μικρή χώρα μέλος η Επιτροπή ΕΚΟΝ επεξεργάζεται την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό του 2014. Ο δε συγητής μας κύριος Λάνγκεν έχει ήδη συντάξει την έκθεσή του και την υπέβαλε τον Οκτώβριο. Συζητείτε δε αυτή. Θέματα ανταγωνισμού λοιπόν θα βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια διάταξή μας και μέχρι τέλους του έτους. Έτσι λοιπόν, στο όνομα της Επιτροπής Οικονομικών ε, Θεμάτων, σας ευχαριστώ για την προσήλωσή σας ε, στην συζήτηση ε, μαζί μας. Αναμένουμε μια σύντομη τοποθέτησή σας της τάξης των 10 έως 15 λεπτών και μετά θα λάβουν το λόγο τα μέλη ανά όπου θα μπορούν τα μέλη να υποβάλουν σύντομες ερωτήσεις και ελπίζω να λαμβάνουν σύντομες απαντήσεις, ερωτήσεις απαντήσεις και βεβαίως αν κάποιος θέσει μια μακροσκελή ερώτηση και λάβει μια εξίσου μακροσκελή απάντηση τα 5 λεπτά έχουν φύγει. Έτσι λοιπόν πρώτα ε, η Επίτροπος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε πρώτα απ' όλα. Είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Και είναι καλό που μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί πιστεύω ότι έτσι έχουμε ένα πραγματικό διάλογο, κάτι το οποίο με βοηθάει και εμένα να έχω νέες ιδέες. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πριν από ένα χρόνο, περίπου ακριβώς ένα χρόνο, αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι μια καλή στιγμή για να προσθέσουμε ένα νέο κεφάλαιο στην συνεργασία μας. Τη Επιτροπή σα με μένα δηλαδή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν για το σχέδιο εκθεσή του όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νομίζω προφανέ να διαβάσετε την έκθεση σε βάθο το βλέπετε ότι πολλά μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Είναι πολλά υποσχόμενη λοιπόν αυτή η συνεργασία. πολύ υποσχόμενη και για τους πολίτες, οι οποίοι έτσι βλέπουν ότι συνεργαζόμαστε προκειμένου να εφαρμόσουμε το δίκαιο του ανταγωνισμού. Η ενιαία αγορά βέβαια αποτελεί και το πετράδι της κορώνας, ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει να προσφέρει η Ευρώπη σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθεί να ισχύει, να είναι ανοιχτή και να λειτουργεί καλά. Και αυτό ακριβώς είναι και ο κοινό μας στόχος. Πιστεύω επίσης ότι έχουμε συμφωνήσει, συμφωνούμε ότι η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι που θα βοηθήσει να πετύχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε επιχείρηση, κάθε εταιρεία πρέπει να έχει την ευκαιρία να λειτουργεί και να κάνει το εμπορικό της όνειρο πραγματικότητα. Δεν πρέπει να εμποδίζεται από μεγάλες επιχειρήσεις, από εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν δεσπόζουσα θέση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή. Οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι υπάρχει ίση μεταχείριση, ότι υπάρχει δικαιοσύνη και ότι έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβαση στην αγορά. Είναι κάτι που το κάνουμε για τους πολίτες, το κάνουμε για τους καταναλωτές. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, τότε και οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και αναπτύσσονται μέσω των προϊόντων τους, μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θέλει κανείς να έχει εμπορικέ δραστηριότητε στην Ευρώπη. Είναι κάτι πάνω στο οποίο έχουμε συμφωνήσει όλοι και αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε την πρωτοβουλία μου προκειμένου να δώσουμε νέα όθηση στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Μιλάω τώρα για τη διαβούλευση την διαβούλευση που έχουμε προκειμένου οι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού τη Ευρώπη, να μπορούν πιο αποτελεσματικά να εφαρμόσουν του κανόνε για τον ανταγωνισμό όπως είπε και ο κύριος Φέντερ, έστειλα ένα email σε εσά την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να ενημερωθείτε περισσότερο για τις δικές μας ιδέες. Θα σας πω λοιπόν λίγα λόγια επ' αυτού τώρα. Γιατί τώρα πάνω από 10 χρόνια οι εθνικές υπηρεσίες για τον ανταγωνισμό έχουν παίξει ρόλο κλειδί προκειμένου να εφαρμόσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού στις χώρες μέλη. Τις χρειαζόμαστε το χαρτοφυλάκιο αυτό βέβαια έχει πολλές αρμοδιότητες στην ε, Επιτροπή. Παρόλα αυτά είναι αναγκαία η συνεργασία μας με τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά μέσω του δικτύου ανταγωνισμού και από το 2004 και μετά έχουμε εγκρίνει πάνω από χίλιες αποφάσεις ε, κατά το μονοπώλιο Antitrust. Οι χώρες ε, μέλη όμως πήραν 85% από αυτές τις αποφάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που δείχνει πώς οι εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να συνεργαστούν καλά υπέρ των πολιτών μας και προς όφελος των πολιτών μας και των καταναλωτών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δικιά του την πλευρά μας εθάρρυνε πάντα να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Αυτοδίκτυο Ανταγωνισμού για πολλούς και διάφορους λόγους. Αν θέλουμε ο ανταγωνισμός να κάνει τη διαφορά στη ζωή των πολιτών μας, Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αρχές μπορούν να παίξουν πλήρως το δικό τους ρόλο. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για τις διαδικασίες ή για τους κανόνες, πρόκειται για την ίδια τη δικαιοσύνη, την ε, ίση μεταχείριση. Οι κανόνες του ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από το σε ποιο κρατό μέλο βρισκόμαστε, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί μερικέ φορέ εφαρμόζεται διαφορετικά. Το ξέρουμε ότι οι επιχειρήσει έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά πρόστιμα ανάλογα με το σε ποια χώρα που βρίσκονται. Μπορεί να είναι από μη μέχρι 25 φορές παραπάνω, αν υπάρχει κάποια παράβαση. Εξαρτάται από το ποια αρχή θα είναι υπεύθυνη και την υπόθεσή τους. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες καταφέρουν να ξεφύγουν από τα πρόστιμα αλλάζοντας το νομικό τους πρόσωπο. Έπειτα, όλες οι εθνικές αρχές δεν έχουν εξίσου τα μέσα για να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους. Είναι κάποιες εθνικές αρχές που λένε ότι θα μπορούσαν να τα καταφέρουν πολύ περισσότερο αν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή τους, αν είχαν περισσότερη ισχύ. Αυτό είναι πολύ βασικό δεν φτάνουν οι κατευθυντήριες γραμμές ή οι ανακοινώσεις. Είμαι πεπισμένη ότι δεν φτάνουν από μόνα τους αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς και ανέλαβα την προηγούμενη εβδομάδα την πρωτοβουλία να αρχίσω να δουλεύω για να καταλήξουμε σε μια νέα νομοθετική πρόταση. Την τελευταία χρονιά οι υπηρεσίε μου ε, κατέγραψαν την κατάσταση πως έχει, συζήτησαν με τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, με τους Υπουργούς, τις χώρες μέλη. Και το υλικό που συλλέξαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εντοπίσουμε πού ακριβώ βρίσκονται τα προβλήματα και τι είδους δράση από την πλευρά μας χρειάζεται για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και στις 4 Νοεμβρίου άρχισε και η δημόσια διαβούλευση. Στόχος της είναι να συγκεντρώσουμε τις απόψει όλων των πλευρών ώστε να αποφασίσουμε τι δράση πρέπει να αναλάβουμε στη συνέχεια. Τρει τομεί μας απασχολούν ιδιαίτερα. Πρώτον, να δούμε τι εγγύσει υπάρχουν ότι οι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού έχουν τα μέσα και του πόρου που χρειάζονται για να κάνουν το δουλειά του. Δεύτερον, ότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να εντοπίσουν και να επιβάλλουν κυρώσει στην περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσει των κανόνων του ανταγωνισμού. Και τρίτον, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι προγράμματα επικούς ε, μεταχείρισης ε, μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο αποτελεσματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν προσπαθούμε βέβαια εδώ να αλλάξουμε την οτροπία των χωρών μελών ή να πούμε εμείς ποια αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό και την εφαρμογή των κανόνων. Όχι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουν όλες οι αρχές στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό λαμβάνοντας υπόψη τι διαφορέ από χώρα σε χώρα, αλλά και από την άλλη μεριά να μην εξαρτάται το αποτέλεσμα από το σε ποια χώρα ζεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να σα ενημερώσω ακριβώ για αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Είναι σημαντικό συγχρόνως να μιλήσουμε και για τη δικιά σα εμπλοκή, εφόσον εσείς είσαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών είναι προφανές ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν που έχω αναλάβει έχει, θέλει να χρησιμοποιήσει το Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης εφόσον ε, βέβαια το επιτρέπει και το περιεχόμενο της ε, πρότασης. Πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε τι μπορεί να πετύχει πολιτική ανταγωνισμό όταν αυτή εφαρμόζεται σωστά και ανεξάρτητα. Είναι πολύ σημαντικό. Οι πολίτες το βλέπουν κάτι σημαντικό και καταλαβαίνουν ότι έτσι γίνεται σωστή δουλειά. Τι εννοώ, εννοώ βέβαια τις αποφάσεις που πήραμε για τις δύο πρώτες περιπτώσεις όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις. Γιατί είπαμε ότι η Fiat τελικά έπαιρνε παράνομα κρατικές ε, επιδοτήσεις από το Λουξεμβούργο και Starbucks από την Ολλανδία. Επαναλαμβάνω ότι αυτές οι δύο αποφάσεις για τις δύο αυτές επιχειρήσεις δίνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τις χώρες μέλη αλλά και προς τις επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για μεγάλες είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για μεγάλες χώρες είτε πρόκειται για μικρές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς το φορολογικό σύστημα για να προσφέρεις τελικά κρατικές επιδοτήσεις. Θέλω επίση να ξεκαθαρίσω ότι Πρόκειται για την αρχή της δουλειά μου, του έργου. Τέλος. Θα συνεχίσω να εξετάζω περιπτώσεις φορολογικών ρυθμίσεων. Αν έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τους κανόνες ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, δεν εφαρμόστηκαν σωστά, θα το κάνω. Και βέβαια, αν ανοιχτεί μια τέτοια υπόθεση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να έχουμε συμπεράσματα. Φροντίζοντας βέβαια πάντα την ποιότητα της δουλειά μα. Συγχρόνως προχωρούμε και αναλύοντας ε, την προσέγγιση μα όσον αφορά τι ε, φορολογικές ρυθμίσει όλε τι χώρε μέλη. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και να δουλέψουμε πως πραγματικέ κατευθυντήριε γραμμές για το πότε οι φορολογικές ρυθμίσει αποτελούν ε, κρατική επιδότηση και πότε αυτή είναι παράνομη. Έχουμε μια κοινή οπτική από όπου και αν προερχόμαστε. Έχουμε μια νέα αγορά, άρα χρειάζεται ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη και αυτό είναι που πρέπει να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους σε όλες τις χώρες μέλη. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούν οι πολίτες να αντιληφθούν το ωφέλη της ε, ενιαίας αγοράς. Και έτσι θα το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν μια δουλειά, θέλουν να φτιάξουν μια επιχείρηση, να καινοτομήσουν και να ενημερώσουν τους πελάτες τους γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ε, σίγουρα θα με ρωτήσετε για πολύ περισσότερα θέματα από αυτά που ανέφερα εγώ και το ελπίζω. Εγώ θα σταματήσω εδώ και να ξέρετε ότι ό,τι μου πείτε θα περάσει και στους συνεργάτες μου. Σας ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όπως είπα και πριν, εκτιμούμε το έργο σας και δίκιο έχετε όταν λέτε ότι η ενιαία αγορά δεν χρειάζεται μονάχα κανόνες ενιαίας αγοράς, χρειάζεται και κανόνες και αποφάσεις για τον ανταγωνισμό. Νέο κεφάλαιο αυτό τώρα των κρατικών επιδοτήσεων μέσω της φορολογίας. Το έχετε ανοίξει και θα συνεχίσετε και εσείς και εμείς να ασχολούμαστε με αυτό. Θα ακολουθήσουμε τώρα το σύστημα DEHONT για να δώσουμε το λόγο στις διάφορες πολιτικές ομάδες με πρώτο το Λαϊκό Κόμμα και τον κύριο Μπάλτς. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Θα ρίξω ιδιαίτερο βάρος στον πρώτο αυτό γύρο σε φορολογικά θέματα. Γιατί για τους περισσότερους εξημών εδώ στην Επιτροπή έχουν κρίσιμη σημασία επί του παρόντος. Έχουμε και αυτή την ειδική επιτροπή για τα φορολογικά. Θα ήθελα να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις. Πρώτα, ποια είναι η θέση σας σχετικά με το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός συστήματος συμψηφισμού όπου θα εξετάζονται οι αποφάσεις tax ruling στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το εάν έχουν ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες μέλη. Έχετε εξετάσει ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα στην πράξη ή οι παρενέργειες ενός τέτοιου συστήματος. Δεύτερο, πρόσφατα ανακοινώσατε δύο αποφασίσεις σχετικά με τα tax ruling. Άρα έχετε ήδη εμπειρία στον τομέα αυτό. ποιο, σε ποιο χρόνο υπολογίζεται να εγκριθούν οι κατευθυντές γραμμές για τις ρυθμίσεις αυτές έτσι ώστε να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και για τις χώρες και για τις επιχειρήσεις. Αυτά είναι η δεύτερη ερώτησή μου λοιπόν. Η απάντηση. Πρώτη ερώτηση για αυτό το κέντρο συμψηφισμού, clearing house. Η απάντηση είναι δεν γνωρίζω. Υπάρχουν και υπέρ και κατά. Ένα από τα κατά είναι ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και να δώσει το αίσθημα στις χώρες μέλη ότι δεν είναι αυτές υπεύθυνε για τα tax ruling που εκδίδουν. Θα πρέπει να είμαστε πλέον φιλόδοξοι, να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα tax ruling δεν θα είναι εργαλείο που να προσφέρει ε, συλλογικά πλεονεκτήματα, αλλά να εξασφαλίζει μια ασφάλεια δικαίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ζητήσουμε και από τον ΩΣΑ και για την ε, ε, διάβρωση της φορολογικής βάσης και για τις αποφάσεις κλπ. Και να περάσουμε σε ένα αυτόματο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για tax ruling και αυτό να γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και περισσότερη διαφάνεια πάνω σε μια κοινή φορολογική βάση. Στη συζήτηση για αυτό το κέντρο συμψηφισμού, και τώρα έρχομαι στο δεύτερο ερώτημά σας, θα έχει σημασία και γι' αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου θα χρειαστούμε πολύ χρόνο για να φτιάξουμε παραδοσιακές, ας το πω έτσι, κατευθυντήρες γραμμές. Γι' αυτό το ερώτημα είναι πόσο σύντομα μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στις χώρες μέλη που να είναι πιο light, αλλά παρόλα αυτά να επιτρέπουν στις χώρες μέλη να δουν πώς μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες μας πλέον διαφανείς και να συμμορφώνονται πλήρως με τις κατευθύνσεις γραμμές για τις κρατικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις με τις αποφάσεις που έχουμε λάβει και αυτές που θα έλθουν ακόμα και με την ανάλυση των tax ruling που έχουμε από τις χώρες μέλη, εκείνες δηλαδή που ακολουθούν το σύστημα αυτό, μπορούμε να τα προωθήσουμε ακόμα περισσότερο για να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις μέσα σε ένα ορατό μέλλον. Σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό σας μείνει ακόμη κύριε Μπάλτς. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Πέτρα Σίμων. Θα τα πω στα γερμανικά εγώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Συγχαρητήρια για τις αποφάσεις σας της προηγουμένης εβδομάδος που δείξατε ότι δεν μιλούμε μονάχα για αθέμητες συμπεριφορές αλλά και για πραγματικά παράνομες συμπεριφορές. Πολλοί είπαν ότι α, αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι παράνομες με την διαπίστωση όμως και εφόσον αυτή ενισχυθεί, αποδείχνεται ότι είναι παράνομες συμπεριφορές αυτές. Όμως οι αποφάσεις αυτές που λήφθηκαν και στην βάση των εγγράφων που διαθέτετε και που λάβατε, είστε σε θέση να εξετάσετε το πλήθος των ενδεχόμενων αυτών περιπτώσεων. Δεύτερη ερώτηση. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Το Συμβούλιο προωθεί τώρα τον εξοπλισμό με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπουν την άντληση κάποιων στατιστικών συμπερασμάτων, αλλά εσείς ως θεματοφύλακες των συνθήκων δεν λαμβάνετε τις προφορίες εκείνες που θα σας έδιναν τη δυνατότητα να παίξετε το ρόλο σας και να εξετάσετε, να ελέγξετε εάν τα tax ruling, οι αποφάσεις τύπου tax ruling, όντως συμμορφώνονται με το πρωτογενές δίκαιο. Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε λοιπόν εσείς ως ελάχιστο ποσοστό για να, ως ελάχιστο ποσό μάλλον, για να μπορείτε να παίξετε τον ρόλο του θεματοφύλακα των Συνδικών. Τρίτο, ο ρόλος της Κομισιόν στην ομάδα Code of Conduct. Έγιναν κάποια προδημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο, τώρα το Σαββατοκύριακο, που δίνουν κάποιες υποφορίε τις οποίες δεν διαθέτουμε εμείς, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν τις διαθέτουμε διότι για λόγους εμπιστευτικότητας οι χώρες μέλη δεν μας διαθέτουν ορισμένα έγγραφα που διαθέτει η ομάδα Code of Conduct. Και τα δημοσιεύματα στον τύπο, στο γερμανικό τύπο, λένε ότι ήδη από χρόνια μέμφονται ορισμένες χώρε μέλη, άλλε για την στάση τους στα tax ruling η Κομισιόν είναι μέσα στο, στην ομάδα Code of Conduct, του κώδικα διοντολογίας δηλαδή. Και αυτή η ομάδα κώδικα διοντολογίας δεν είναι ανεξάρτητο όργανο που να μην μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε λοιπόν υποχρέωση εσείς ως θυματοφύλαξη των συνθήκων, εφόσον λάβετε πληροφορίες μέσα στην ομάδα του κώδικα διοντολογίας, θα πρέπει η Γενική Σας Διεύθυνση να τις ανακοινώσει πληροφορίες αυτές και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το έμεσο ερώτημά μου. On uh, Για το πρώτο ερώτημα, για το αν ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε αρκετά. Καταρχήν, δεν ε, θέλω εγώ να μετατραπώ στην Ευρωπαϊκή Αρχή, Φορολογική Αρχή, γιατί έχουμε κρατικές φορολογικές αρχές, αλλά είναι και θέμα απόρων. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι βεβαίως να εξασφαλίσουμε ότι από εδώ και στο εξή θα έχουμε tax rulings που θα είναι απόλυτα σύμμορφα με τις ε, αρχές και την νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, πιστεύω με την καθοδήγηση από, με βάση αυτές τις υποθέσεις που είχαμε μέχρι στιγμής. Εδώ λοιπόν σαφώς βλέπουμε τι συμβαίνει και δίνουμε μια μεθοδολογία μέσω των αποφάσεων μας για το πώς θα επανυπολογιστούν ο φορολογικός φόρτος των τριών αυτών εταιριών. Αλλά βασικά αυτό απασχολεί και τον ΟΣΑ, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσουμε όταν κάνουμε εσωτερική τιμολόγηση ότι υπάρχει σχέση λόγος ένα προς ένα σε σχέση με τις τιμές αγοράς, έτσι ώστε οι εσωτερικές τιμές να μην είναι ο τρόπος για να μεταφέρονται κέρδη σε περιοχές χαμηλής ή ε, καθόλου φορολογίας. Και αυτό νομίζω το σύστημα, αν χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο, νομίζω πως μπορούμε έτσι με αναπερίπτωση να έχουμε τόσο πολλές ε, καθοδήγηση ε, που ποτέ θα το ελπίζαμε. Να μην χρειαστεί δηλαδή να επαναλάβουμε τα όσα κάνουν οι εθνικές αρχές. Για το θέμα τώρα της στατιστικής. Εγώ δεν γνωρίζω την θέση του συναδέλφου Μοσχοβησή που έχει ευρύτερα την ευθύνη για την φορολογία. Αλλά για μας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ βοηθητικό το ότι έχουμε ισχυρά μέσα ώστε να μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε στη διάθεσή μας. Και όπως γνωρίζετε, όταν συζητούσαμε το αίτημα για ενημέρωση περί tax ruling από όλα τα κρατημέλη, είπαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, όλο ένα και καλύτερα εργαλεία για να μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Έχουμε λοιπόν τώρα τα κατάλληλα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας και δεύτερον ε, χρησιμοποιούνται ε, για το, τώρα, για την ομάδα του κώδικα διοντολογίας. Είναι πολύ χρήσιμο τόσα κάνουν, πιστεύω. Είναι δύσκολο να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να πούμε ότι τα όσα συζητώνται εκεί θα πρέπει να μπουν στη δουλειά μας, διότι πιστεύω ότι η ομάδα του κώδικα διοντολογίας έχει στην ουσία προετοιμάσει το έδαφος για μια αλλαγή στο πώς βλέπουμε την εταιρική φορολόγηση και βρίσκω το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ επικοδομητικό. Σας, δίνω κάποια... Σας έδωσα λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, αλλά πρέπει να προσέχουμε τους κανόνες. Ο κύριος Σταμπάτη, εξ ονόματος της ομάδας ECR. Εγώ Μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Σπίλμπορν που δεν μπορεί να παρακολουθήσει την σημερινή μας συνεδρίαση διότι χρειάστηκε να πάει την κόρη τη επιγόντως στο νοσοκομείο. Επίτροπε, καταρχήν θα σας συγχαρώ για το πρόσφατο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο και ε, η Ολλανδία προσέφεραν συγκεκριμένα ε, ωφέλη, φορολογικά ωφέλη στην ε, Starbucks την Fiat με τη... παρανόμως. Ε, θα πρέπει λοιπόν επίσης να σας συγχαρώ για το ότι δείξατε μια ισχυρή βούληση ώστε να τεθεί τέλος σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τώρα έχω δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μου πείτε σε πώς και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως οι δύο αποφάσεις της ε, Κομισιόν θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη και στις εταιρείε. Επίσης θα ήθελα να να γνωρίζω ποια είναι η αξιολόγησή σας για τις πρόσφατες επιτυχείς συμφωνίες ε, του ΟΣΑ που βασίζονται, που βασίζονται στο σύμφωνο για την ε, για, την εταιρική φορολόγηση και για την απογόρευση μεταφορών κερδών, καθώς και για το θέμα της αλλαγής έδρας. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις στη φορολόγηση. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση και αν ναι, σε ποιο βαθμό βλέπετε ότι η διάβρωση του, της, βάσης, της φορολογικής βάσης αλλά και η μεταφορά κερδών θα βοηθήσουν στο να προωθηθεί ένα κείμενο για ολοκληρωμενη φορολογική, ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη φορολογική βάση, όπως ξέρετε ότι προτείνουν αρκετά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. I, hope that... Καταρχήν, ε, καταρχάς πιστεύω ότι η, συν, η κόρη συναδέλφου θα γίνει καλά γρήγορα. Ε, να σας πω τώρα Πιστεύω ότι το αποτρεπτικό στοιχείο είναι αρκετά ισχυρό και αυτό το έχω τονίσει από την πρώτη μέρα όταν, υπέβαλα, όταν παρουσίασα τις δύο αποφάσεις. Ότι δηλαδή εδώ υπάρχει ένα μήνυμα για τα κρατημέλη και για τις εταιρείε. Αυτό που αντί να πούμε ακριβώς αυτό το ποσό θέλουμε να, να μπορέσουμε να συλλέξουμε. Εμείς προτείναμε μια μεθοδολογία ώστε να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Τώρα για το project του ΟΣΑ για την διάβρωση τη βάση και τη μεταφορά κερδών. Το εκτιμώ πολύ και ελπίζω πως θα εγκριθεί και από τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όταν συνεδριάσουν γιατί δείχνει ακριβώς ότι αυτό ε, το πρόβλημα είναι ευρύτερο από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε όλο ένα και περισσότεροι να συμφωνήσουν σε αυτό και να εξασφαλίσουμε ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου ε, υπάρχει και δημιουργείται το κέρδο. Έχω ήδη μάθει βέβαια ότι πρέπει κανείς πολύ να προσέχει με, όταν χρησιμοποιεί πολύ ισχυρή, πολύ έντονη γλώσσα, αλλά εάν εφαρμοστεί σωστά είναι πάρα πολύ καλό μέσο για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Τρίτον, αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό εταιρικό χώρο φορολόγησης, εγώ πιστεύω πως όχι. Και αυτό δεν έχει κάνει μόνο με τις ε, εθνικές, αλλά και με μικρότερες εταιρείε μπορεί να έχουν ε, θηκατρικες σε τρία κράτη-μέλη, ας πούμε και θα πρέπει να γνωρίζουν έτσι πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογική βάση και θα μπορούν ίσως να εξοικονομήσουν ε, τα χρήματα ε, που θα δίναν σε φοροτεχνικούς ε, ή λογιστές κτλ. Και κάπως τα πράγματα να είναι πιο απλά, αν και αυτή είναι πολύ μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά τη φορολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να σβήσετε το μικρόφωνο σας παρακαλώ κύριε Σταμπάτη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εξ ονόματος των φιλελευθέρων, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόζα Ιβάντσες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέστε γερμανικά ο κύριος Σαμονές. Συνεχίστε αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θέλω να μου πείτε περισσότερα για τη Starbucks και την Fiat. Ελπίζω να προχωρήσετε περισσότερο σε βάθος. Έχω δύο ερωτήσεις τώρα. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Μπογκελεγό. Χαίρομαι για την έσταση μετά από πέντε χρόνια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει και να τελειώσει τη δουλειά αυτή από τα Android σε άλλους τομείς. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν νέα για το τι γίνεται με αυτό το θέμα. Τώρα για τα πρόστιμα από την Google έχω καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βάση για να επιβάλλει πρόστιμα. Η Microsoft είπε το ίδιο πριν από μερικά χρόνια. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτά. Τα πρόστιμα θα υπολογίζονται ανά έτος ζημιάς. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να τα υπολογίζουμε από το 2006. Από τότε άρχισε η ζημιά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή η χρονιά αυτή, όχι. Τώρα, όσον αφορά τον ανταγωνισμό στις αεροπορικές εταιρείες. Και εδώ θα έπρεπε να προσέξουμε πιο πολύ τις κρατικές ενισχύσεις. Με τον 868 του 2004 όσον αφορά τις ε, τιμές, είδαμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν ήταν αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει ότι τέτοιες ενισχύσεις κανονικά είναι παράνομες αν πάνε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Οπότε ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να έχει και μια ρήτρα ε, θεμητού ανταγωνισμού και όσον αφορά τις εξωτερικές μας σχέσεις στην αεροπλοεία. Και οι κανόνες όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των αεροπορικών εταιριών κριτήρια ελέγχου θα έπρεπε να τα αναθεωρήσουμε όσον αφορά το πακέτο αεροπλοίας. Πρώτα απ' όλα, να σας απαντήσω όσον αφορά την Google και πώς έχουν και τα πράγματα. Η έρευνα για τα Android άρχισε τον Απρίλιο και είμαστε στη μέση της διαδικασίας, οπότε δεν μπορώ να σας πω πότε θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η Google επίσης απάντησε στις ενστάσεις μας το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία ευαίσθητα στην απάντηση, τα αναλύουμε και θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία και από την Google και από τρίτα μέρη. Αυτό ακριβώς θα ζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Για το θέμα των προστήμων τώρα. Τα πρόστιμα καθορίζονται βάσει της διάρκειας και της σοβαρότητας της παράβασης. Και μπορεί να είναι και πολύ βαριά τα πρόστιμα, γιατί ακριβώ θέλουμε να δρουν αποτρεπτικά. Άρα, όταν πρόκειται για καρτέλ δεν είναι ε, ένα ακόμα πρόστιμο, όχι, πρέπει να αντικατοπτρίζει και τη ζημιά την οποία έχει προκαλέσει το καρτέλ η δεσπόζουσα θέση. Πρόσφατα επιβάλαμε πρόστιμα σε διάφορες εταιρείες με καρτέλ το οποίο είχαν επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά στα οπτικά σου οπτικές Οι 160 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν απατώμε. Οπότε ναι, βάζουμε πρόστιμα σε επιχειρήσεις εάν έχουν προκαλέσει ζημιά στην ευρωπαϊκή αγορά. Όσον αφορά τώρα την αεροπλοία. Αυτό που λέτε το έχουμε ήδη κάνει. Με την DG Move, τη Γενική Διεύθυνση Move δηλαδή, συνεργαζόμαστε διότι έχουμε βρεθεί σε διάφορες περιπτώσεις που υπάρχει σύνδεση διαφόρων υποθέσεων, κάτι το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλούς πολίτες. Δεν πρόκειται δηλαδή για τον ανταγωνισμό μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός συνεργάζομαι με τον συνάδελφο Μπούλς που επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτούς τους τομείς όταν θα έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αεροπλοεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ από την ΚΟΕ. Η Παλώμα Λόπες Μπερμέο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ισπανικά θα υποβάλω την ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως στην πολιτική ανταγωνισμού είναι ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να ρυθμίζει μια αγορά η οποία να λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών και όχι υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι το εργαλείο αυτό πρέπει να είναι χρήσιμο για να διορθώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς και να διασφαλίσει ότι θα τηρούνται όλες οι ευρωπαϊκές διατάξεις. Όσον αφορά τη ρύθμιση τώρα για την λειτουργία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις σας και ναι, συμφωνώ με αυτά που λέτε. Αλλά εξακολουθώ να ανησυχώ για το πώς θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των οργάνων αυτών, ανεξαρτησία απέναντι στις χώρες, τις ίδιες, αλλά και απέναντι στις ίδιες τις αγορές που πολλές φορές παρεμβαίνουν στην νομοθετική διαδικασία. Έχω και τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις τέλος. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να αντιμετωπίσει το κοινωνικό dumping, το οποίο λαμβάνει χώρο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αν ναι, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Θα υιοθετηθούν ε, μέτρα για τη Starbucks και την Fiat ώστε τα ποσά τα οποία θα επιστραφούν να επιστραφούν στις χώρες όπου παράχθηκε η αξία αρχικά. Δεύτερον, όσον αφορά τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία, με τα νέα νομοθετικά μέτρα έχουμε τεράστιες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτού τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα να απαντήσω στο πώς οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν να δρουν ανεξάρτητα. Αυτός είναι ένας τομέας σχετικά με τον οποίο έχουμε διάφορε ιδέε, αλλά γι' αυτό θέλουμε και την δημόσια διαβούλευση, γιατί μπορεί να επιτεθεί η ανεξαρτησία αυτή με πολλού και διαφορετικού τρόπου. Και γίνεται ήδη με πολλού και διαφορετικού τρόπου σε διάφορε χώρε. Πάει πάρα πολύ καλά η ανεξαρτησία αυτή. Αλλού υπάρχουν περιθώρια βελτίωση ακόμα. Και εννοείται ότι θα θέλαμε στη δημόσια διαβούλευση να έρθει κόσμο και να μα πει να, εκεί και εκεί πάει στραβά και θα θέλαμε να διορθωθεί αυτό και αυτό. Δεύτερον, για το κοινωνικό ντάμπινγκ. είναι μάλλον θέμα των συναδέλφων και όχι τόσο δικό μου, αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε νέους κανόνες που λένε ότι δεν μπορεί κανείς να προσφέρει στήριξη σε μια επιχείρηση να πάει σε μια χώρα εάν θα χαθούν οι ίδιες, ε, ο ίδιος αριθμός ε, θέσεων απασχόλησης ε, από τη χώρα προέλευσης. Το θέμα δεν είναι να έχεις κάποιο κέρδος. Μπορεί να μην έχει άμεσα σχέση με το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο δείχνει ότι μας απασχολεί το γιατί γίνεται αυτό που γίνεται και όχι για στραβούς λόγους, για λόγους ενισχύσεων. Η τρίτη σας ερώτηση είχε να κάνει με την επιστροφή των ε, ποσών που εισπράχτηκαν ε, παράνομα στις χώρες όπου παράχθηκε η αξία. Δεν είναι δικό μας θέμα να το αποφασίσουμε εμείς. Εμείς ε, φροντίζουμε να επιστραφούν τα ποσά τα οποία δόθηκαν ως ενισχύσεις παράνομα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και δεν θα ξαναπώ καν πώς θα γίνει, γιατί πραγματικά πώς να βρούμε ένα τέτοιο μέτρο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν έτσι όπως λέτε. Είναι όμως μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει ευρύτερα και όχι μόνο όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τη φορολογία. Γιατί έχει να κάνει με πολύ περισσότερα ζητήματα. Τέλος, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν γνωρίζω πολύ καλά την ισπανική περίπτωση, θα επανέλθω. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας να συμπεριληφθούν στους ενεργειακούς πόρους αυτούς καθ' αυτούς. Είτε πρόκειται για την ηλιακή, είτε πρόκειται για την νεολική, Ξέρετε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και ότι πράγματι μπορεί να πετύχει αυτό που λέμε και να είναι και πιο φτηνό και για τους καταναλωτές. Αλλά για την ισπανική περίπτωση θα πρέπει να επανέλθω αργότερα γιατί δεν έχω υπόψη μου περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Εκ μέρου των Πρασίνων, ο Φιλίπ Λάμπερτ τώρα έχει το λόγο. Επίτροπε, όταν ε, με ρωτά κανείς για την Επιτροπή Γιούνκερ, έχω κάποια καλά πράγματα να πάω, αλλά εσείς είστε η λαμπρή εξαίρεση και είμαι σοβαρός για αυτά που λέτε. Εγώ, είμαι, ε, εγώ ε, θέλω να καταγραφεί αυτό για το τι κάνετε πρέπει να σας συγχαρώ ε, για τους πολίτες. Ο, ο κάτοχός σας, ο Αλμούνια, άνοιξε το, αυτό το ταμπού, αλλά εσείς ε, συνεχίζετε με μεγάλο ενθουσιασμό. Είπατε ότι δεν είναι το τέλος αυτό, θα διερευνήσετε, είπατε και άλλε υποθέσεις. Υπάρχουν χιλιάδε rulings τέτοιου είδους, αποφάσεις τέτοιου είδους. Πώς θα τις επιλέξετε και πώς θα εντοπίσετε ποιες υποθέσεις θέλετε να, να ξαναερευνήσετε, γιατί έχετε περιορισμένου πόρους στη διάθεσή σα, όπω και όλοι μα. Ε, δεύτερη ερώτηση, Volkswagen. Σε πολλέ χώρε η εταιρεία ή οι πελάτες που αγοράζουν ε, προϊόντα από αυτή την εταιρεία έχουν λάβει επιδοτήσεις επί τη βάση ε, λανθασμένων ε, πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί στρέβλωση της αγοράς. Πώς θα προχωρήσετε λοιπόν αν φανεί ότι όντως η Volkswagen έκανε απάτη, αυτό το ξέρουμε, αλλά μετά και τα κράτη ε, αν πήραν ε, παράνομα χρήματα από τη Volkswagen για να αγοράσουν στην ουσία μη πράσινα αυτοκίνητα. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Ε, πραγματικά ε, με συγκινούν. Δεύτερον, ε, έχετε δει και υπάρχουν πάρα πολλά rulings. Τώρα αναλύουμε 300 από κράτη-μέλη τα οποία κάνουν τέτοιες ε, συμφωνίες, tax rulings. Έχουμε παραδείγματα όπου είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, δεν έχουμε να ρωτήσουμε και λεπτομέρειες και μετά βρίσκουμε ε, ποιες είναι οι υποθέσεις οι οποίες είναι οι πιο προφανείς. Κατάφορες. Γιατί πιστεύω και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη ότι εκεί ίσως θα έχουμε καλύτερα, ε, καλύτερη εμπειρία και θα αποκομίσουμε διδάγματα όλοι και οι επιχειρήσεις και εμείς. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από, μια, από κάποια πλευρά γιατί αν έχουμε κάποια αμφιβολία για το ότι αυτά τα, αυτές οι αποφάσεις δεν ακολουθήθηκαν σωστά, θα πρέπει να ε, κάνουμε διώξεις με τους πόρους που έχουμε. Όσο γίνεται οργανωνόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα πυρήνα εργαζομένων που ασχολούνται με αυτό το θέμα αλλά βεβαίως όπως είπατε όλοι είναι υπό την πίεση των περιορισμένων πόρων ωστόσο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη Volkswagen. Η υπόθεση αυτή είναι ακόμα υπό εξέταση, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τι θα προκύψει τους επόμενους μήνες. Οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει η Volkswagen ήταν ξεκάθαρες, έχουν μπει μέσα στην έρευνα, στην ανάπτυξη και τέτοιου είδους πράγματα, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω ένα ποσό, ένα σύνολο για το πόσα χρήματα δηλαδή έχουν λάβει οι κρατικές ενισχύσεις, έχει λάβει η Volkswagen. Κάτι το οποίο όμως είναι ξεκάθαρο είναι ότι από την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους κάθε κράτος μέλος ε, θα δημοσιεύει τι κρατικές ενισχύσεις δίνει και σε ποιους. Αυτό ήταν μέρος του προγράμματος για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Και επίσης η αποκέντρωση των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Στο μέλλον λοιπόν θα μπορεί κανείς να δει ποιο κράτος δίνει ποια κρατική ενίσχυση σε ποια εταιρεία. Ε, νομίζω πως αυτό θα διευκολύνει την κατάσταση αν προκύψουν άλλου τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ναι, αλλά εσείς θα ζητήσετε να επιστραφούν αυτές ε, οι κρατικές ενισχύσεις, θα το εξετάσετε. Ε, αυτή η Volkswagen πήρε ενισχύσεις για να πουλήσει πράσινα αυτοκίνητα δεν, εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο Μάρκο Βάλλη από το FTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι σήμερα εδώ και απαντά στα ερωτήματά μας και πρέπει να πω την αλήθεια ότι καθόλου δεν σας ζηλεύω σε αυτή την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή γιατί υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά ξεσπάνε σκάνδαλα και απαιτείται δικαιοσύνη για τα θέματα της φορολογίας γιατί εγώ γυρίζω όλη την Ιταλία ας πούμε και εξηγώ υποθέσεις όπως αυτή της Fiat και της Starbucks στους πολίτες και φυσικά και θα θέλαν πιο συγκεκριμένε απαντήσει από τα κρατημέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει κάπως να συμφωνήσουν γιατί είναι παράλογο. Αν και τιμωρείται ας πούμε μια πολυεθνική όπως η Fiat και η Starbucks, αυτές μετά πηγαίνουν και πληρώνουν ακριβώς στις χώρες όπου τις διευκόλυναν και που ζημίωσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και οι πολίτες ρωτών πότε θα έχουμε πραγματικά ένα σύστημα φορολογικό συνεπές το οποίο δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνο των πολυεθνικών. Θα ήθελα πραγματικά να μπορέσουμε σε κάποια χρόνια να μπορέσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις αυτές. Είναι ευπρόσδεκτες και οι δημόσιες διαβουλεύσεις λοιπόν για την εξέβρεση συστημάτων για τη συνεργασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν θα πρέπει να βάζουμε μόνο κείμενα επιτάπητος για να λέμε ναι κάτι κάνουμε και τελικά να μην ολοκληρώνεται κάτι. Υπάρχει κάποιος οδικό χάρτης, υπάρχει μια πραγματική βούληση γιατί κάθε φορά που λαμβάνεται μια απόφαση σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ Βλέπουμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, υπάρχει δυνατότητα για να μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών διαφάνεια που θα μπλοκάρει αυτό το σύστημα, αλλά τελικά τα κράτη-μέλη ε, συνεχίζουν να δρουν ε, κατά το δοκούν. Ε, οι πολίτες πρέπει να πιστεύουν τους θεσμούς ή απλώς μας κοροϊδεύουν και μας κοροϊδεύουν και τα κράτη μας ε, με τη σειρά τους. Εγώ είμαι 30 χρονών ε, μόνο, αλλά από τότε που έχω αρχίσει να προσπαθώ ε, βλέπω πως είναι δύσκολα τα πράγματα. αλλά δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου με πράγματα που ενώ μάλλον προωθούνται κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον. Η Επίτροπος τα σχόλιά σας με καθιστούν αισιόδοξοι. Όσο περισσότερο στοχεύουν οι πολίτες, δηλαδή εντοπίζουν το ενδιαφέρον τους στο θέμα αυτό, τόσο περισσότερο μπορούμε να προχωρήσουμε. Τίποτε δεν εμποδίζει τις χώρες μέλη να αλλάξουν και να αρχίσουν να αλλάζουν ήδη από σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πραγματικά λόγος, υπάρχει καθήκον των ψηφοφόρων να επιμείνουν ώστε να μπουν τα πράγματα αυτά στην ατζέντα των κυβερνήσεων. Τα πράγματα, εφόσον δηλαδή χρησιμοποιούν tax ruling, να γίνονται σε συμμόρφωση με το ε, τεθειμένο δίκαιο. Και εφόσον εργαστούμε όλοι μαζί, κανείς δεν θα αισθάνεται ότι δεν υπάρχει πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού και ότι η... κάποια επιχείρηση μπορεί να αποφύγει την φορολόγηση. Είναι σημαντικά αυτά, διότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και στις κρατικές ενισχύσεις με την ομοθεσία. Τα πράγματα αυτά περάσουν τώρα βεβαίω με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, αλλά να αρχίσουν οι χώρες μέλη να προχωρήσουν δηλαδή σε αλλαγές, αυτό μπορεί να γίνει ήδη αμέσως. Και γι' αυτό εγώ προσπαθώ να προχωρήσω όσο γίνεται γρηγορότερα. Να δώσω δηλαδή κατευθύνσει για το πώ μπορούν να γίνουν τα πράγματα αυτά, εφόσον οι χώρε μέλη έχουν αμφιβολίε για το πώ να χειριστούν το θέμα, διότι συμφωνώ μαζί σα, Αισθάνομαι και εγώ ότι οι άνθρωποι περιμένουν από εμά να αλλάξουμε το σύστημα, διότι βλέπουν χιλιάδε επιχειρήσεων που πληρώνουν κανονικά του φόρου του Και υπάρχουν άλλε επιχειρήσει που έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφεύγουν και ορισμένες από αυτές μάλιστα με πολύ επιθετικό τρόπο. Και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι έχουν αντιληφθεί ποια μέτρα, ποια βαριά μέτρα έλαβαν οι κυβερνήσεις για να εξηγιάνουν τους προϋπολογισμούς. Η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα υπόσχεται πολλά και νομίζω ότι όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως κάνει η δική σας Επιτροπή Τάξε, τόσο καλύτερο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Φέρμπερ. Από άλλη ε, πολιτική ομάδα δεν βλέπω άλλο συνάδελφο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, κύριο Λάνγκεν. Ευχαριστώ και, και εγώ και εσάς κυρία Επίτροπε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την καλή συνεργασία, συνεργασία μαζί σας. Έρχομαι σε δύο θέματα. Πρώτο, οι αποφάσεις tax ruling. Εμένα μου φαίνεται παράξενο το εξής μια απόφαση δηλαδή. Οι ποινές που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις πηγαίνουν τελικώς όμως στις χώρες που δεν είναι τα θύματα, αλλά οι δράστες. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Είναι οι χώρες οι οποίες πρόσφεραν αυτά τα φορολογικά πλονεκτήματα και τελικώς αυτές πράττουν. Αυτό ίσως να τις καθησυχάζει, αλλά είναι τα ίδια πράγματα όπως με τις ποινές για τα καρτέλ. Οι ποινέ για τα καρτέλ όμω πηγαίνουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι οι ποινέ θα πρέπει να λάβουν την ιδία οδό όπω οι ποινέ, οι χρηματικέ ποινέ δηλαδή, που επιβάλλονται για ε, υποθέσει καρτέλ. Διότι τα θύματα είναι άλλε χώρε μέλη, οι οποίες ε, επιχειρήσει των οποίων δηλαδή δεν έχουν απολαύσει αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με εκπλήττει τώρα το γεγονό ότι κάτω χώρε και οι και το Λουξεμβούργο λαμβάνουν τώρα τα χρήματα αυτά, διότι μπορούν να πούν Α, δεν φταίει εμεί, φταίει η κακιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, ορισμένε απειλούν με προσφυγέ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει θεμελιωδώ αυτό, έτσι ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη πίεση για εθελούσιε αλλαγέ βεβαίω στι χώρε μέλη. Δεύτερο, για την πρότασή σα για την συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ Ανταγωνισμού. Η πρότασή σας μου φαίνεται όρθη και αυτή εφόσον είναι σωστή ανάλυση που κάνω, αναφέρεται ιδίω στι συνεργασίε με στόχο δημιουργία καρτέλ. Μιλήσατε για παραπάνω από χίλιε υποθέσει, όπου απέδωσε και έχουν γίνει έρευνε για υποθέσει καρτέλ. Αυτό είναι σωστό. Τα κενά εκεί πάλι εντοπίζονται στι κρατικέ ενισχύσει. Από τα πολλά χρόνια που είμαι ευρωβουλευτή και τι πολλέ συζητήσει που έχω διεξαγάγει για τι κρατικέ ενισχύσει από τι εθνικέ αρχέ. Εκεί δεν είναι αρμόδιες οι εθνικές αρχές καρτέλ, αντικαρτέλ δηλαδή, αλλά οι κυβερνήσει των χωρών μελών που αυτές δίνουν τι κρατικέ ενισχύσει. Και μέχρι τώρα λοιπόν η συνεργασία αυτή δεν έχει αποδώσει, γι' αυτό η ερώτησή μου έχει ως εξή. Πώς βλέπετε αυτό τον τομέα της συνεργασίας, δεν χρειάζεται εδώ να ασκηθεί η μεγαλύτερη πίεση της χώρε μέλη. απάντηση της Επιτρόπου Βεστάγκερ. Από τη δική μου σκοπιά, τα χρήματα που ανακτούν οι φορολογικές αρχές καταλήγουν στους φορολογούμενους. Έχετε δίκιο βέβαια που λέτε ότι είναι παράδοξο ότι δηλαδή η χώρα που χορήγησε αυτό το selective advantage εισπράττει τελικώ τα χρήματα. Αυτό ισχύει βέβαια για κάθε περίπτωση κρατικής ενισχύσεως και ε, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω πώς να δημιουργήσω ένα σύστημα που να λέει ότι πάει στην τάδε χώρα ή στην δίνα χώρα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σχετικά με, τα, με το ποια κέρδη αποκομίζουν οι επιχειρήσεις και πώς φορολογούνται αυτά στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτά βέβαια με την φορολογική βάση του ε, φόρου επιτεριών. Όπως το βλέπω εγώ όμως οι φορολογούμενοι των χωρών ε, ανακτούν τελικά τα χρήματα. Δεύτερο, έχετε δίκιο όταν λέτε σχετικά με τις ερωτήσεις που θέτουμε στις ε, εθνικές αρχές του κυρίως έχουν σχέση με υποθέσεις καρτέλ. μπορούν να λάβουν περισσότερες αποφάσεις οι κυβερνήσεις για, για θέματα κρατικών ενισχύσεων οι πολιτική προϋποθέσεις να είναι διαφανείς και να εξηγήσουν τους πολίτες με ποιο τρόπο πανούν τα χρήματα. Αυτό θα είναι αποτελεσματικό με την έννοια ότι αν η χώρα μέλος εγκρίνει την ε, κρατική ενίσχυση, αυτή θα γίνεται σωστά. Αυτό νομίζω ότι είναι και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διερευνήσει Κάποια φορά και αυτεπαγγέλτος, εάν υπάρχει περίπτωση παράνομης κρατικής ενισχύσεως σε κάποια χώρα μέλος. Και είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό. Αυτό θα πρέπει να το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες οι διαδοχικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές να το εξετάζουν. Διότι είναι ζήτημα ανταγωνισμού εφόσον μια μεγάλη ή πλούσια χώρα μέλος μπορεί να προσφέρει φορολογικά πλεονεκτήματα σε ορισμένες επιχειρήσεις στην ουσία να τρέπει την ισοτιμία στους όρους του ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, την Μπορσάνη. Ναι, ορίστε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Πολύ θα ήθελα να έχω τις απαντήσεις σας στη συνέχεια και όλα αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν από τα συμπεράσματα της Επιτροπής για τις Φορολογικές Ρυθμίσεις. Ό,τι έκανε μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις παρατηρήσεις, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Μέχρι τώρα Έχουμε μιλήσει για μεγάλα ψάρια που αρνούνται να πληρώσουν φόρους, αλλά οι δικές σας υπηρεσίες σίγουρα θα πάνε περισσότερο σε βάθος για να βρούνε εκτός από αυτά τα μεγάλα ψάρια και τα μεσαία ψάρια που εποφελούνται από φορολογικές ε, ρυθμίσεις διευκόλυνσης. Θέλω να επιστήσω στην προσοχή σας ένα θέμα που είναι από τη χώρα μου η Ουγγρική κυβέρνηση πρώτα απ' όλα κατάργησε πλήρως τον τζόγο. Και μετά ως παραχώρηση τέδωσε έναν μόνο. Αυτός ο ένας όμως έτσι μπορεί να επωφεληθεί με τέτοιες ρυθμίσεις. Είναι βέβαια ένας φίλος του Πρωθυπουργού. Πήρε αυτή τη διευκόλυνση γιατί, γιατί η κυβέρνηση έκανε ένα νόμο ε, με τον οποίο χρησιμοποίησε τον όρο availability, ότι μόνο αυτός υπήρχε. Κάτι άλλο τώρα, πιο γρήγορα, γιατί απαντήσατε πολλές φορές σχετικά με αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για το πρόσφατο φαινόμενο ε, υποθέσεων που βρίσκονται σε διάφορες χώρες και που σε ορισμένες χώρες απαγορεύονται κάποιες δραστηριότητες, σε κάποιες άλλες δεν απαγορεύονται. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Πρώτα απ' όλα, το θέμα του μεγέθους του ψαριού όπως το θέσατε είναι βέβαια ένα ζήτημα. Εμείς ασχοληθήκαμε με ένα μέρος της Starbucks, της Fiat και γι' αυτό και η ανάκτηση των χρημάτων είναι κάπου ανάμεσα σε 20 με 30 εκατομμύρια σε σχέση με ολόκληρη τη Starbucks δεν είναι μεγάλο το ποσό. Σε σχέση με ολόκληρη τη Fiat δεν είναι μεγάλο το ποσό. Πάντως το σημαντικό εδώ είναι το θέμα της αρχής. Ότι δηλαδή πρέπει να φροντίσεις, να πληρώσεις και να ξέρεις ότι υπάρχουν όρια για το πόσο μπορείς να πληρώσεις πριν πούμε ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνεις. Το βασικό δηλαδή είναι το θέμα της αρχής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι επόμενες περιπτώσεις είναι κάπως διαφορετικές, αλλά έχουν να κάνουν με τη φορολογία και θα πούμε περισσότερο όταν θα έχουμε καταλήξει. Τώρα για το τζόγο στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε ρωτήσει διάφορα ζητήματα, αλλά ευχαριστώ να επανέλθω, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις με τις Ουγγρικές Αρχές, έχουμε ρωτήσει για την φορολόγηση των εθνικών και των ξένων επιχειρήσεων. Όσον αφορά, τώρα, όσον το sharing. Εδώ με τη συνάδελφο Μικόφσκα συνεργαζόμαστε για την ενιαγορά αγορά, ακόμα και για τις μεταφορές, διότι είναι αλήθεια ότι είναι διαφορετικά τα χαρτοφυλάκια, αλλά όταν συνεργαζόμαστε τότε αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα πώς λειτουργούν αυτές οι επιμερισμένες υπηρεσίες κοινέ υπηρεσίες. Οι ψηφιακέ επιχειρήσεις δημιουργούν κάτι νέο, κάτι που προσφέρει νέες δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους. Εμείς είναι απόλυτα θεμητό να ρωτάμε για την φορολογία, για την ασφάλεια και αυτό ακριβώ κάνουμε αυτή την εποχή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρου του ΕΛΚ, η κυρία Χάνοβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ χαίρομαι που είσαστε εδώ στην Επιτροπή μας και συγχαρητήρια για το μέχρι τώρα έργο σας. Χρειάζεται πολύ ενέργεια αλλά και θάρρος για να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις σοβαρές περιπτώσεις όπως αντιμετωπίσατε εσείς. Η ερώτησή μου θυμίζει λίγο αυτό που ακούσαμε από τον προλαλήσαντα. Την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσατε ότι η ψηφιακή μας ε, οικονομία πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν ψηφιακά από άλλες χώρες χωρίς πρόβλημα. Το έχουμε πει αυτό εδώ και καιρό βέβαια. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα οι καταναλωτές σε τέτοιες αγορές. Η ψηφιακή οικονομία όμως μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και όσον αφορά τα προϊόντα και όσον αφορά τις υπηρεσίες χωρίς να υπάρχουν ε, στρεβλώσεις. Αλλά παρόλο που ξέρουμε πόσο πολύ προς το συμφέρον της οικονομίας μας θα ήταν κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά τίθενται πολλά ζητήματα ανταγωνισμού όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες αγορές. Οπότε ε, ευχαριστώ πολύ για τις έρευνες που κάνετε όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμετες πρακτικές. Ρωτάω όμως, υπάρχει τρόπος, εντάξει μπορώ να το πηγαίνω πολύ μακριά, αλλά όσον αφορά τη στρατηγική για την ενιαία αγορά που ξεκίνησε πρόσφατα και για την ατζέντα όσον αφορά την ε, οικονομία αυτή μέσω συνεργασίας, εσείς αυτή την έρευνα θα τη χρησιμοποιήσετε σαν βάση για να προχωρήσει περισσότερο το εμπόριο αυτό. Επίτροπο, Ελπίζω. Πραγματικά ελπίζω. Γιατί βέβαια όταν κάνουμε μια τέτοια έρευνα την κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Κάτω από 10% των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων κάνουν διασυνοριακά ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι περίεργο, γιατί θα, πρέπει να είναι πιο εύκολο κανονικά, αντί να αναγκάζονται να έχουν ένα κατάστημα στην άλλη χώρα κλπ. Οπότε προσπαθούμε να δούμε γιατί. Είναι θέμα ε, συμβάσεων, είναι θέμα το ότι δεν ποδίζουν οι προμηθευτές, για ποιο λόγο. Προσπαθούμε λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο και να ενημερώσουμε και τους συναδέρφους, γενικά εκείνους που έχουν περισσότερες νομοθετικές αρμοδιότητες, ώστε όταν θα αναλύσουμε τις ε, απαντήσεις που θα πάρουμε, και ευχαριστώ πολύ και για σας, να χρησιμοποιήσουμε τις απαντήσεις αυτές. Ο αντιπρόεδρος Σάντσεπ, για παράδειγμα, εκείνος μπορεί να φροντίσει να προωθήσει περισσότερο τη διευκόλυνση αυτή. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό για όλους μας και για τον ανταγωνισμό, αυτό καθε αυτό, να ενημερωθούμε για τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι, λοιπόν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενος για τους σοσιαλιστές, η κυρία Γκίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η αλληγουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την όθηση της οικονομίας και την απασχόληση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Συμβάλλει δε με 35 με 45 δις στο ΑΕΠ της χώρας μας ετησίως. Είναι εξαιρετικά σημαντική ιδέα η χαλιβουργία στη δική μου περιφέρεια και νομίζω ότι στη δική μου μόνο περιφέρεια πρόκειται για 500.000, μάλλον 250.000 κόσμο που απασχολείται. Το πρόβλημα το βασικό είναι το ψηλό κόστος της ενέργειας. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην περιφέρειά μου που έχει μπει σε διαδικασία πτώχευσης ονομάζεται Καπάρο και μάλιστα Σήμερα το πρωί ε, ο γενικός διοικητής της ε, πέθανε, υποτίθεται επειδή αυτοκτόνησε. Όμως εκατοντάδες χιλιάδες ε, θέσεις απασχόληση εξαρτάται από αυτό την εταιρεία. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός Αρμόδιος, ο κ. Ντάβιντ, κατά κατηγορεί την Ένωση ότι δεν έχει δράσει και αυτό, οφείλεται αυτή η κατάσταση στις κρατικές ενισχύσεις και ότι δεν έχει γίνει τίποτα ε, στα θέματα κατά του ντάμπινγκ. Γι' αυτό το λόγο είπε ότι έχουμε κρίση, επειδή πέφτει δηλαδή διαρκώς η τιμή του χάλιβα. Και ορισμένες φορές ε, ε, έχουμε λόγο να δώσουμε κρατικές ενισχύσεις. Η Κομισιόν έχει κάνει εξαιρέσει ε, στο παρελθόν σε άλλου τομεί. Έχει επιτρέψει δηλαδή κρατικέ ενισχύσει σε περιπτώσει ανάγκη. Εδώ θα δώσετε τη δυνατότητα αυτή και θα οριστικοποιήσετε το, ε, τους όρους του αντι έναντι του φθηνού χάλιβα που εισάγεται στην Ένωση. Νομίζω ότι η χαλιβουργία είναι σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη. Σε πολλά κρατημέλη έχουμε σημαντική χαλιβουργία και βέβαια έχουμε πολλά προϊόντα που ε, ε, κατευθύνονται στην κατασκευαστικό τομέα. Η Ευρώπη ε, εξακολουθεί δε να είναι εξαγωγέας χάλιβα προς τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό είναι ε, δείγμα της ποιότητας του χάλιβα που παράγεται στην Ευρώπη. Κάτι επίσης που έμαθα είναι ότι υπάρχει με τεράστια ποικιλία χαλιβουργικών προϊόντων. Οπότε αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με το dumping έχουν πολύ δύσκολη δουλειά για να μπορέσουν να κάνουν ε, ε, τη δουλειά που πρέπει, όταν δηλαδή βλέπουν ότι εισάγεται χαμηλότερες τιμές χάλιβας, αλλά ε, να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα ότι ε, εισάγεται ο χάλιβας που χρειάζεται στα στις κατάλληλες τιμές. Από όσο γνωρίζω, ο αρμόδιος τομέας ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα αντι-dumping, κατά του dumping, ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία των ευρωπαϊκών ε, χαλιβουργιών. Επίσης, έχουν ληφθεί, έχει ληφθεί απόφαση από τους επικεφαλείς κρατών το 2013 και που δεν επιτρέπει να δίνεται ε, κρατική ενίσχυση στην χαλιβουργία είχαν γίνει οι αναλύσεις πριν να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις από τα κράτη-μέλη. Αυτό βεβαίως που κάνουμε είναι ότι συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος για εξαιρέσεις όταν πρόκειται για τους ε, μεγάλους καταναλωτές ενέργειας να ας πούμε όπως οι κανόνες για τη μετάβαση σε ανανεώσιμη οικονομία αυτοί οι κανόνες να χρησιμοποιούνται με όσο γίνεται διαφανέστερο τρόπο και συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ιδέες με βάση τις δικές του ιδέες τη στιγμή που μιλάμε ώστε αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν να μπορέσουν να χρησιμεύσουν και για το Ηνωμένο Βασίλειο όπως έχουν χρησιμεύσει και για άλλα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, και εδώ, τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπάλτσε, εξενόματος του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η μία αφορά την, ε, τις αναφορές αναχώρα. Επίτροπε, πιστεύετε ότι ορισμένα είδη ε, τέτοιων αναφορών αναχώρα θα χρησιμοποιηθούν ώστε να εντοπιστούν οι παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις πολυεθνικές στο μέλλον και θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μην τοποθετηθούν εταιρείε σε μειονεκτική θέση ε, έναντι των εκτός ένωσης αντιπάλων τους ή ανταγωνιστών τους. Δεύτερη ερώτηση αφορά πιο συγκεκριμένο θέμα του προπολογισμού για το 2016. Η Επιτροπή μας στην γνωμοδότησή της για τον προπολογισμό του 2016 προτείνει τη χορήγηση περισσότερων πόρων για τις δαπάνες που σχετίζονται με την πολιτική ανταγωνισμού ώστε να προχωρήσει ο αγώνας κατά του επιθετικού φορολογικού προγραμματισμού των πολυεθνικών εταιριών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση όσον αφορά την ανάγκη επιπλέον πόρων. Ευχαριστώ. Για τις αναφορές αναχώρα. Πιστεύω πως αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν πριν να μπορέσει να υποβάλει κάποια πρόταση η Κομισιόν. Νομίζω πως είναι ενδιαφέρον που ήδη θεωρείται ότι η έκθεση, οι αναφορές αναχώρα αφορούν τον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Σημαίνει δηλαδή ότι αν μπορούν να τα καταφέρουν και σιγά σιγά αρχίζουν να ευημερούν, υπάρχει χώρος για τις αναφορές αναχώρα χωρίς αυτό να είναι επιβλαβές ε, για τις εταιρείες ή ζημιογόνο για τις εταιρείες. Δεν νομίζω ότι αυτέ οι αναφορέ μπορούν να δείξουν ε, τι παράνομε κρατικές ενισχύσει. Εκεί πρέπει να μπει κανεί στι λεπτομέρειε για να, ε, να εξετάσει τα συγκεκριμένα tax rulings. Αλλά μπορεί να αποδείσουν ε, τι παράνομε κρατικές ενισχύσει, Γιατί πόσο έχουμε αναχώρα αναφορέ είναι πιο προφανέ ότι που πληρώνει κανεί του φόρου του. Αν του πληρώνει δηλαδή εκεί που έχει και την έδρα του και που δημιουργείται το κέρδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δουλέψουμε προ αυτή την κατεύθυνση η Δεύτερο είναι το, για να απαντήσω στην ερώτησή σα, πώ να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μην ε, ζημιωθούν ή να μην βρεθούν σε μηνυκτική θέση επειδή είναι εντάξει. Δεν έχω ακόμα την απάντηση σε αυτό. Με του συναδέλφου. εργαζόμαστε από αυτού, γιατί θα πρέπει να είναι Να, να, να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη διαφάνεια. Βέβαια το θέμα είναι την άλλη σας ερώτηση με τους πόρους είναι γεγονός ότι πάντα μπορείς να χρησιμοποιήσεις περισσότερους πόρους. Το θέμα είναι πόσους περισσότερους. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη συνάδελφο που διαπραγματεύεται τον προπολογισμό για το 2016 με εσά και άλλους συναδέλφους και θα θεωρήσω το αποτέλεσμα ως κάτι το δεδομένο και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με όποιους σπόρους θα έχω για να εξακολουθήσω να επιδιώκω αυτό αυτούς τους κοινού μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα εξ ονόματος των σοσιαλιστών, ο συνάδελφος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ισπανικά θα μιλήσω. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, διαδικαστικά. Έχουμε κάποια ημερομηνία για να ξέρουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για την Apple και την Amazon. Δεύτερον, μετά από αυτά που είπε και η Νίνα Γκίλ, γίνεται ευρεία συζήτηση για την δυνατότητα η Κίνα να θεωρηθεί οικονομία αγοράς. Εσείς έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε θεμητό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά και άλλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι καταλαβαίνω, εμπλέκονται στο θέμα του διεθνούς εμπορίου. Θέλω όμως να ξέρω τη δικιά σας την άποψη. Πιστεύετε ότι μία οικονομία η οποία, στην οποία το καθεστώς επηρεάζει την παραγωγή μπορεί να θεωρηθεί οικονομία αγοράς τη στιγμή που η Κίνα εξορισμού είναι κατευθυνόμενη η οικονομία. Ο όγκος των εισαγωγών χωρών που δεν τηρούν την οικονομία αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα να κορυδεύουμε τους αυτούς μας. Τι βάση είναι αυτή για τον θεμητό ανταγωνισμό στην Ευρώπη στο μέλλον. Θέλω τη γνώμη σας από αυτού. Η Επίτροπος. Δεν μπορώ να σας δώσω μια ημερομηνία για αποφάσεις όσον αφορά τις υποθέσεις Apple και Amazon. Η Amazon εξάλλου ξεκίνησε αργότερα ως υπόθεση για μας, ως έρευνα από την Apple. Δεν μπορώ να σας δώσω ημερομηνίες γιατί δεν έχω ημερομηνίες. Όλα θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία που έχουμε, από τα στοιχεία που θα συλλέξουμε, γιατί συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Όσον αφορά την Κίνα τώρα. Επίσημα, αν θεωρηθεί η οικονομία της αγοράς σε Κίνα, έχει κάποιες επιπτώσεις βάσει και του ΠΟΕ. Από όσο γνωρίζω λοιπόν, πρέπει να συνετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αποφασίσουμε να θεωρήσουμε την Κίνα σαν μια οικονομία αγοράς όπως οποιαδήποτε άλλη οικονομία αγοράς. Πάντως μπορεί κανείς να είναι οικονομία αγοράς με διαφορετικούς τρόπους. Η Ευρώπη είναι οικονομία αγοράς παρόλο που σε ένα βαθμό είναι ρυθμισμένη η αγορά αυτή. Ε, ρυθμίζεται η εργασία, ρυθμίζονται και άλλα. Είναι μια ρυθμισμένη οικονομία. Ας αφήσουμε τον ε, ΠΟΕ και τον ορισμό για αργότερα. Πάντως συνεργαζόμαστε με την Κίνα και έχουμε μάλιστα υπογράψει ένα έγγραφο εργασίας προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των ε, συγχωνεύσεων και αν κοινοποιηθεί κάτι τέτοιο σε περισσότερο από μία νομολογία θα το εξετάσουμε. Η Κίνα θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ό,τι διαφορές και αν έχουμε, πάντως είναι καλό να συντονιζόμαστε, γιατί έτσι μπορούμε να εφαρμόζουμε ε, κανόνες ανταγωνισμού μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Και είναι σημαντικό αυτό, παρόλο που βέβαια ο ορισμός, οι διαδικασίες που ισχύουν μπορεί να διαφέρουν. Πρέπει πάντως να συνεργαζόμαστε με την Κίνα ώστε να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση για το πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις δικές μας χώρες. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τέλος ο εισηγητής μας, ο εισηγητής της ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Επανέρχομαι σε μια φράση που είπατε στην πρώτη σας απάντηση ότι τα χρήματα επιστρέφονται στους φορολογούμενους. Δεν θίγονται όμως οι φορολογούμενοι του Λουξεμβούργου αλλά άλλοι όπου δημιουργούνται τα κέρδη. Εγώ νομίζω ότι εδώ ε, υπάρχει ένα λογικό σφάλμα όταν τα χρήματα δηλαδή επιστρέφονται στο Λουξεμβούργο που έχουν ένα χιλιοστό του ΑΕΠ της Ευρώπης και ακόμα ε, ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολλά φορολογικά έσοδα για άλλους λόγους. Είναι πολύ διαφορετική γνώμη μου, να είστε σίγουροι. Τώρα, πώς, μπορείτε, πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντονότερα στην δημοσίευση οδηγιών, κατευθυντηρίων γραμμών, κατευθύνσεων για παράδειγμα για τη συμμετοχή των αρχών ανταγωνισμού. Και τρίτο, σε μια μονάχα υπόθεση περιφερειακού χαρακτήρα στις 4 Νοεμβρίου η Κομισιόν έδωσε μια γνωμοδότηση για μια υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον Nürburgring. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα και δεν έχει απαντηθεί ποτέ από την Κομισιόν εάν η διαδικασία ήταν ουδέτερη, και, ουδέτερη για τον ανταγωνισμό δηλαδή και διαφανής. Οι προσφεύγοντες λένε ότι δεν ήταν διαφανής ούτε ουδέτερη η ε, υπόθεση αυτή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προσωπικά, αλλά η αξιωματούχη της δεν έχει επιληφθεί. Ε, εγώ γνωρίζω την ιστορία αυτή και δεν κατανοώ καθόλου την επιχειρηματολογία των συνηγόρων. Η Επίτροπος το γεγονός ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουδέτερο και ανεξάρτητο είναι νομίζω από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Και να μην μιλήσω καν για τους δικούς μας ελέγχους που έχουμε, τα λεγόμενα checks and balances, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι υποθέσεις αυτές όντως έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό ένα προφανό, προφανές σημείο αφιτηρίας όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει περισσότερη άμεση ευθύνη είναι με τους φορείς, τους εθνικούς φορείς και αρχές ανταγωνισμού. Θα πράξω πάντα το δυνατό για να διασφαλίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι συνομοθέτης στην πρόταση αυτή. Βέβαια, μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα στην δημόσια διαβούλευση και να αλλάξει αυτό. Αλλά ο στόχος με αυτός είναι διότι νομίζω ότι θα ενισχυθεί η εργασία αυτή με τον τρόπο αυτό και το αποτέλεσμα θα είναι βελτιωμένο, εάν δηλαδή συμμετάσχει το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης. Βεβαίω χρειάζεται πρόταση για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αν δεν ακούσαμε τίποτα που να είναι ιδιαίτερα ανατρεπτικό στη δημόσια διαβούλευση, αυτό νομίζω είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Και όσον αφορά την προηγούμενη πρόταση όπου ήταν συνομοθέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία κατέληξε πολύ καλά. Έτσι, θεωρώ ότι είναι σωστό να κάνουμε το προφανές και τα πρώτα πράγματα να γίνουν πρώτα. Δεύτερο, για τη φορολόγηση και την ανάκτηση. Ευχαριστώ να το συζητήσω σε ευρύτερη βάση από τις κρατικές μόνο ενισχύσεις. Είναι προφανέ είδα εγώ του κανονισμού όταν πρόκειται για θέματα κρατικών ενισχύσεων, η ανάκτηση των ενισχύσεων έτσι γίνεται. Και έχει εγκριθεί πριν από καιρό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Χρειάζεται μια άλλη συζήτηση να γίνει, ειδικά για τη φορολόγηση, που να έχει ευρύτερη οπτική και να συμμετάσχουν περισσότεροι συναδελφοί από τη δική πλευρά και από τη δική μας. Ο πρόεδρος Φέρμπερ, σας ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσαμε την, ε, τον κατάλογο των απολυτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Στην αρχική σας τοποθέτηση είπατε πολύ ευγενώς ότι ε, αναμένετε να μάθετε πράγματα από εμά και να εμπνευστείτε, αλλά εμείς μάθαμε πολλά από σας, άρα ήταν καλό αυτό το δούνε και λαβήν. Η επόμενη ανταλλαγή πληροφοριών μα θα είναι στις αρχές του επομένου Ετου πλέον. Ελπίζω να έχει επιτευχθεί πρόοδο σε πολλούς από τους τομεί που μνημονεύσαμε σήμερα και στους οποίους εργάζεστε για την ώρα. Οι λεπτομέρειες για την έκθεση για τον ανταγωνισμό, για την πολιτική ανταγωνισμού, το σχέδιο κατατέθηκε στις 13 Οκτωβρίου. Την 5η θα διεξαχθεί συζήτηση και εξέταση τροπολογιών. Η ψηφοφορία προβλέπεται να γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή. Στην δε Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταλήξει στις 18 Πρώτου 2016. Αυτό είναι ο σχεδιασμός για την ώρα για να εγκριθεί. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί λοιπόν τότε. Δι, διακόπτεται εδώ η σημερινή μα συνεδρίαση και αρχίζουμε αύριο ε, το πρωί τη 9 η ώρα με το περίφημο θέμα των MIFID.